Ολοκληρώθηκε λοιπόν τώρα αυτή η συζήτηση και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τώρα θα έχουμε μία δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Και γι' αυτό τον ο, ο Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, πάντοτε πριν τα Χριστούγεννα συζητούμε για τα παιχνίδια. Και σωστό είναι γιατί είναι η εποχή όπου ως επιτοπλίστων ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για τα παιχνίδια και είμαι ευγνώμων που γίνεται η συζήτηση πάλι εφέτος γιατί η ασφάλεια των παιχνιδιών είναι μία αέγνια από κοινού του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και του Συμβουλίου και όπου έχουμε τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πύχη. Η συζήτηση σήμερα το απόγευμα προκλήθηκε και από διάφορα άρθρα στις εφημερίδες ε, σε ένα κράτος μέρος και δεδομένα εις ε, την Γερμανία από ένα Ινστιτούτο για την έρευνα και διερεύνηση των κινδύνων και την εποπτεία και αυτοί δεν απευθύνθηκαν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε η γερμανική κυβέρνηση απευθύνθηκε κατευθείαν εις ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε απλώς ότι δηλώσεις έγιναν στον τύπο και τι διαβάζεται στο γερμανικό, σε γερμανικές εφημερίδες. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να συζητήσουμε συζητήσουμε ακόμη και αν συζητείτε μέχρι τούδε μόνο μέσω των εφημερίδων. Η ανάλυση των εκθέσεων μας αποδεικνύουν ότι υπάρχουν τέσσερα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Καταρχήν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ εύκολο να απαντηθεί διότι σύμφωνα με δηλώσεις της Γερμανικής Εποπτικής Αρχής υπάρχουν ε, παιχνίδια που κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά και εξετάστηκαν και βρέθησαν να μην ε, ε, καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθετία. Όταν λοιπόν ένα κράτος διαπιστώνει κάτι τέτοιο είναι υποχρεωμένο να αποσύρει αμέσω όλα τα παιχνίδια, να ειδοποιήσει την Επιτροπή, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά τρόπον ώστε όλα τα προϊόντα παντού στην Ευρώπη να αποσυρθούν αμέσω και να υπάρξει μία άμεση απαγόρευση ε, ε, εισαγωγή εάν προέρχονται από εκτός Ευρώπης. Ελπίζω ότι με το ΑΠΕΞ θα σταλούν τα οι αναγκαίες ανακοινώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και γι' αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα δεχθεί και θα προσυπογράψει ε, όλα αυτά τα μέτρα. Μέχρι στιγμή όμως όπως σας είπα έχουμε μόνο ενημέρωση από τον τύπο. Και πρέπει να σας πω ότι η εποπτεία της αγοράς είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ούτε της Επιτροπής, ούτε του Συμβουλίου, ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη και μόνο ε, νομικά είναι δεσμευμένα και υποχρεωμένα να εξασκούν αυτή την εποπτεία της αγοράς και αν διαβάσω για τη Γερμανία ότι είναι αμφισβητή αμφισβητούμενο εάν η γερμανική εποπτική αρχή παρακολουθεί πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη στην περίπτωση αυτή ε, να ε, απευθυνθεί προς την ε, εποπτική αρχή. Το δεύτερο θέμα είναι επίσης ένα παλιό θέμα το οποίο είχε εξετάσει και συζητήσει διεξοδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οδηγία για τα παιχνίδια και είχε υπάρξει και ονομαστική ψηφοφορία για την ε, υποχρεωτική πιστοποίηση των παιχνιδιών από μία τρίτη αρχή από μια ανεξάρτητη αρχή. Η πρόταση είχε διατυπωθεί από τη Γερμανία, από την υποπτική αρχή. Ε, σωστά απερίφθηκε η, ε, η πρόταση αυτή ε, διότι ανεξάρτητη εποπτική αρχή δεν θα δημιουργούσε καμία επιπρόσθετη ασφάλεια για την κατάσταση των παιχνιδιών και τα παιχνίδια δεν είναι πρωτότυπα όπως ξέρουμε το πρόβλημα μας τα παιχνίδια αυτά είναι εάν σε όλη τη διαδικασία κατασκευής έχουν γίνει σεβαστές από όλους τους ε, ε, εισαγωγεί ή κατασκευαστές των διαφόρων τμήματων οι υποχρεώσεις. Θα έπρεπε λοιπόν ένας κατασκευαστής να φέρει την ευθύνη ασχέτως του που βρίσκεται στον κόσμο για το προϊόν το οποίο θέτει στην αγορά. Εάν λοιπόν υπάρξει αυτή η αξιοπιστία τότε θα πρέπει να συζητήσουμε με τη συγκεκριμένη χώρα να βελτιώσει την παραγωγή της. Και εδώ επί του προκειμένου πει το, ε, το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται για την Κίνα με την οποία συζητάμε και λέμε ότι εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή παιχνιδιών θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι γίνονται ε, μεν ε, βελτιώσεις αλλά πρέπει να διασφαλιστεί ότι ότι σέβονται όλες τις προδιαγραφές μας. Επίσης, η χρήση χημικών ουσιών στα παιχνίδια, ένα πολύ λεπτό θέμα. Το πολιτικό καθήκον το οποίο είχα αναλάβει σαν επίτροπος και αναθέσει στους συνεργάτες μου είναι, είναι πάρα πολύ αυστηρή και η θέση αυτή καλυβόταν και από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή από το 2011 βαθμιαία θα πρέπει να υπάρξουν οριακές τιμές οι οποίες στην ε, στιγμή της υιοθετήσεως θα πρέπει να καλύπτουν το state of the art, δηλαδή την καλύτερη δυνατή κατάσταση του προϊόντος πράγμα όμως το οποίο ξεπερνέται συνέχεια διότι υπάρχουν νέες ε, διαπιστώσεις και γι' αυτό συνειδητά έχουμε αποφασίσει ότι οι νέες, ε, τα νέα επιτέγματα που διαπιστώνουν ότι ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά τοποθετημένος μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει νομοθεσία πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αξιολογεί τα προϊόντα και είναι απαραίτητη. Δύο ε, κοινοποιήσεις υπήρξαν επί του θέματος αυτού εφέτος καταρχήν μέσω μιας επιστολής της Ομοσπονδιακής Υπουργού Γεωργίας προς τα εμένα και αμέσως ε, ζήτησα να επιληφθεί η ε, Επιστημονική Επιτροπή και αναμένουμε στο πρώτο εξάμεινο του 2010 το αργότερα το, την έκβαση αυτής της εξετάσεως και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν νέες διαπιστώσεις θα πρέπει αμέσως να διατυπώσουμε μία πρόταση να ε, ε, γίνει ακόμη πιο αυστηρή η οδηγία η οποία ακόμη δεν έχει ισχύσει και θα ισχύσει το 2011. Η δεύτερη περίπτωση που είναι κάποιος περίπλοκη και πιο δύσκολη να εξηγηθεί αναφέρεται στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και πρόκειται για ουσίες ε, με τις ε, οποίες ε, ασχολούμαστε όλοι αλλά και εδώ έχουμε ενδείξεις ότι οι οριακές τιμές για αυτά τα, τους πολιτικούς κυκλικούς αρωματικούς ε, ε, υδρογονάνθρακες είναι ίσως πολύ υψηλή. Ε, περιμένουμε και πάλι τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης για να προβούμε σε διορθώσεις. Πρόκειται εδώ για ένα πρόβλημα το οποίο ίσως δεν καταλαβαίνουμε σαν πολιτική. Πρόκειται για τεχνικά θέματα πάρα πολύ περίπλοκα. Και ε, θα έπρεπε να σας πω ότι επειδή πρόκειται για φυσικές παρατηρήσεις πάρα πολύ περίπλοκες εγώ δεν τις καταλαβαίνω και δεν έχω την απέτηση να τις καταλαβαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να πούν ότι έχουν γνώση επί του θέματος. Άρα μέχρι ενός βαθμού εξαρτώμαθα από τους επιστήμονές μας ε, στους οποίους πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη για να μπορέσουν να επιλύσουν το πρόβλημα διότι διαφορετικά ε, θα διαπιστωθεί ότι ε, μία, μία απόφαση επιστημονική δεν ήταν σωστή. Εμείς όμως σαν πολιτικοί είμαστε σε μια δύσκολη θέση μεταξύ της ανθρωπιστικής αντιμετωπίσεως και της επιστημονικής αντιμετωπίσεως. Σαν πολιτικοί έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά στο επάγγελμά μας και γι' αυτό οι ε, κανόνες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις συστάσεις των επιστημονικών ε, επιτροπών. Πρέπει όμως να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι τόσο σοβαρό ώστε η παραμικρή ε, η παραμικρή ε, υπόνοια ότι μπορεί να υπάρξουν ε, νέες διαπιστώσεις θα πρέπει να εξετάσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προωθείτε στους Και το τελευταίο θέμα είναι ενοχλητικό διότι άκουσα από ένα Ινστιτούτο ενός κράτους μέλους που θα έπρεπε τουλάχιστον να σέβεται τις εκατότατες προδιαγραφές ε, ότι ε, ε, για ελαστικά όπου υπάρχει, υπάρχει πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία από ότι για τα παιδιά δεν έχει γίνει σεβαστή και αυτό είναι απαράδεκτο το οποίο και πρέπει να καταγγελθεί διότι υπάρχει υπάρχουν, υπάρχουν κατασκευαστές ελαστικών οι οποίοι χρησιμοποιούν έλαια τα οποία προϋπάρχουν από την εποχή του Ρίτς και ε, χρησιμοποιούν οριακές τιμές οι οποίες είναι τεράστιες δηλαδή ε, το εκατονταπλές από αυτές τις οποίες θα έπρεπε να έχουμε και ερχόμαστε εις ε, ορισμένα σημεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου για την χρήση ορισμένων ελαίων και για την κατασκευή ορισμένων ελαστικών θα έπρεπε να έχουμε ίχνοστοιχεία και διαπιστώνουμε ότι ε, ε, δεν, ε, δεν εφαρμόζονται οι επιταγές. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι γι' αυτό τον λόγο υπάρχει μία κατάσταση η οποία ε, ε, δεν επιτρέπει σε κάποιον να διατυπώσει μία έγκυρη γνώμη. Όσον αφορά όμως τη συγκεκριμένη οδηγία έχουμε προσπαθήσει ώστε βάσει των ε, βελτίστων γνώσεών μας να κάνουμε ό,τι είναι ε, δυνατόν καλύτερο. Για να το επιτύχουμε αυτό οι νέες διαπιστώσεις ανα πάσα στιγμή μπορούν να ενσωματωθούν στην νομοθεσία ιδίω όσον αφορά τα παιχνίδια για να μπορεί να, τα παιχνίδια που κατασκευάζονται να καλύπτονται από την ε, ε, καλύτερη δυνατή έρευνα. Τώρα πρώτος ομιλητής για το ΕΛ και έχει ο κύριος Φαμπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την σαφήνεια και την ειλικρίνεια των, ε, ε, των του τον ε, κύριο Επίτροπο και θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και να πω ότι θέλουμε να γνωρίζουμε όλες τις επικίνδυνες ουσίες να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την προστασία της υγείας των παιδιών μας και ιδίως πριν από τα Χριστούγεννα όπως είπα είπατε ε, κύριε Επίτροπε και οι γονείς και οι παππούδες πρέπει να ξέρουν ποια παιχνίδια είναι ασφαλή για τα παιδιά τους και τι παιχνίδια μπορούν να αγοράσουν για τα παιδιά τους. Ε, γι' αυτό και στη Γερμανία θα πρέπει οι αρχές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και ε, γι' αυτό ε, θα πρέπει ε, να ξεπεράσει κανείς και τις, τα πρότυπα του Ρίτς. όσο αφορά τις λεπτομέρειες, θυμάστε ότι σας είχα γράψει μία επιστολή σχετικά με τις επιστημονικές διαπιστώσεις. Σας είχα λοιπόν παρακαλέσει να καλέσετε και άλλους επιστήμονες από τη Γερμανία και ιδίω κτηνιάτρους για να μας ε, ενημερώσουν και να συγκρίνουν ε, τις, ε, τα επίπεδα των ουσιών αυτών στο παρελθόν και τώρα. Και το, η κατάληξη είναι ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθούν. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται απλώς για το μπαλάκι το οποίο τσουλάει ο ένας τον άλλον, αλλά πρόκειται για μία σοβαρή διαμάχη μεταξύ επιστημόνων που διαπιστώνεται σαφώς στη Γερμανία και γι' αυτό κάνω μία έκκληση προς εσάς κύριε Επίτροπε για να μπορέσετε να φέρετε όλα τα επιστημονικά Ινστιτούτα σε μία συνεννόηση για την καλύτερη έκβαση. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ράπτη για δύο λεπτά για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κάθε χρόνο αυτή την εποχή οι γονείς μεσολαβούν για να φτάσουν γράμματα για τα δώρα στον άγιο βασίλη. στα γράμματα αυτά τα παιδιά ζητούν παιχνίδια. ένα από αυτά τα παιχνίδια θα μπορούσε να είναι αυτό εδώ όπως αυτό εδώ θα μπορούσε να είναι ένα από τα 104 παιχνίδια τα οποία ήλεγξε το ομοσπονδιακό γερμανικό ινστιτούτο που είναι αρμόδιο για να δει τους κινδύνους σε σχέση με τα καταναλωτικά αγαθά άκουσα προηγουμένως τον κύριο επίτροπο ουσιαστικά να επιπλήττει το ινστιτούτο το οποίο έκανε τη δουλειά του. τον άκουσα επίσης να ρίχνει ευθύνες στους επιστήμονες. τον άκουσα επίσης να ρίχνει ευθύνες στα κράτη μέλη στα οποία ανήκει η εποπτεία. τα άκουσα όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως άκουσα επίσης ότι συνεχώς μας έλεγε με πολύ ειλικρίνεια και με αδιάσυστα στοιχεία ότι κάθε προηγούμενη οδηγία βελτιώνεται κάθε τόσο με καινούρια στοιχεία και μόνο αυτό το γεγονός πιστοποιεί ότι το ομοσπονδιακό γερμανικό ινστιτούτο έκανε σωστά τη δουλειά του άρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. όσον αφορά δε την οδηγία η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το 2011, για τις χημικές ουσίες ξέρετε ότι θα εφαρμοστεί το 2014. και υπάρχει και κάτι ακόμη στις δεκαεπτά δεκεμβρίου μεθαύριο δηλαδή έρχεται στην επιτροπή το κάθε κράτος μέλος να παρουσιάσει το σχέδιό του σε σχέση με τον κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς. αυτά έχουν άμεση σχέση με τη χριστουγεννιάτικη αγορά αυτά έχουν άμεση σχέση με την υγεία των παιδιών μας που παίζουν με παιχνίδια που εμείς τους αγοράζουμε. και τέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή η συζήτηση για τα παιχνίδια. κανονικά η συζήτηση για τα παιχνίδια και την ασφάλεια πρέπει να γίνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και αυτό είναι ευθύνη της επιτροπής. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενο μιλητής είναι ο κύριο Κρόισμαν για τους φιλελεύθερου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η τοποθέτηση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου σχετικά με τις καρκινογόνες ουσίες βασίζεται σε την αρχή what is reasonable achievable και στηρίζουμε αυτή την άποψη. Επίσης ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εάν οι οριακές τιμές που έχουν καθοριστεί για τα παιχνίδια ε, γίνονται σεβαστές. Ζητάτε επίσης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2011 να μπορέσουν να καθοριστούν οι οριακές τιμές για τα παιχνίδια σε τέτοια επίπεδα ώστε να αποκλείεται οποιοδήποτε κίνδυνος για την υγεία των παιδιών παιδιών. Άλλωστε λέγεται ότι χημικά τα οποία μπορούν να προκαλέξουν καρκίνο ή ε, άλλες βλάβες ε, να μην επιτρέπονται στα προσβάσιμα τμήματα του παιχνιδιού πράγμα το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και δια του σεβασμού των οριακών τιμών. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εποπτεία διότι γενικώ υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών όταν πρόκειται ε, για εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει επιπλέον να ελέγξουμε τα παιχνίδια και να δούμε αν στα εισαγόμενα όντως γίνονται σεβαστές οι οριακές τιμές. Ε, έκτον, εάν είναι σωστό είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε χαμηλότερες προδιαγραφές για παιχνίδια που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι δέχεται οι και υπάρχουν ορισμένες απειλέ να αποκλειστούν μόνο τα δηλητηριώδη παιχνίδια πράγματα οποία είναι ε, αντιπαραγωγικό και δεν επιτρέπει να υπάρξει μια κοινή αγορά. Θα έπρεπε λοιπόν ε, να επέμβει και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Ρούλε τώρα για τους πράσινους χωρίς μικρόφωνο. Ωραία. Τώρα, ε, τώρα ισχύει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία, ε, κύριε Επίτροπε. Ε, ζητήσαμε αυτή τη συζήτηση για να μπορέσει να διευκρινίσει κανείς τι είναι σωστό από τις κατηγορίες και τι είναι απλούστατα λαϊκισμός. Καλό θα ήταν να έχει γίνει πριν φτάσουμε στον τύπο, αλλά ακόμη και σήμερα κάλλιο αργά παρά ποτέ. Χαιρετίζω την ανακοίνωση ότι θέλετε να προσαρμόσετε την νομοθεσία και θα ήθελα να πω ότι οι νέοι καρκίνοι στα παιδιά κάτω των 15 ετών από το 1980 έως το 2006 αυξήθηκε. Ε, υπάρχουν πολύ περισσότεροι όγκοι καρκινογόνοι στα παιδιά και πρέπει να επαγρυπνούμε να δούμε αν οι αριθμοί είναι σωστοί και να αντιδράσουμε και αν η τελευταία μελέτη του Ομοσπονδιακού ο Ινστιτούτου δείχνει ότι ε, δεν φτάνει η οδηγία για την πρόληψη των καρκίνων και των καρκινογόνων ουσιών θα πρέπει να δράσουμε κατά τρόπον ώστε να αποφύγουμε να χρησιμοποιούνται ουσίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν 40 τσιγάρα ε, και κάθε στιγμή είναι σημαντική θα πρέπει να ζητήσουμε από να μπορέσουν να σεβαστούν αυτές τις οριακές τιμές. Είναι και θέμα τιμής, αλλά το θέμα τιμής δεν μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της αγοράς. Αλλά εδώ μιλάμε για παιδιά. Οι πολιτικοί θα πρέπει να επέμβουν, θα πρέπει να αυξήσουμε τις προδιαγραφές και βεβαίως είμαστε, είναι οι εθνικές αρχές υπεύθυνε για την εποπτεία, δεν είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από τη Γερμανία να δραστηριοποιηθεί στο θέμα της εποπτείας αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε περίπτωση αφιβολίας δεν πρέπει να δράσουμε και να προσαρμοστούμε εις ε, την επιστήμη και γι' αυτό ελπίζω ότι σύντομη θα έχουμε μία πρόταση στο Κοινοβούλιο και θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις οριακές τιμές με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Τώρα προχωρούμε στους επόμενους ομιλητές. Πρώτα πρώτα την κυρία Τάισεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ασφάλεια των παιδιών μας που είναι και οι πλέον ευάλωτοι καταναλωτές αποτελεί προτεραιότητα για την ομάδα μου και για όλους εμάς. Θελήσαμε λοιπόν μια εργασία στο δυνατόν αυστηρότερη με ένα σαφέ πλαίσιο και είχαμε πολύ και καλή συνεργασία με του εκπροσώπου τη Προεδρία, του Συμβουλίου, τη Επιτροπή και όλου του συζητητέ, όλου του υπεύθυνου όλων των πολιτικών ομάδων. Κάναμε λοιπόν αρκετά καλή δουλειά και σε πρώτα ανάγνωση καταλήξαμε σε συμφωνία. τα θεσμικά όργανα τότε ήταν πεπισμένα ότι ενέκριναν ε, μια, ένα νομοθέτημα το οποίο ήταν αρκετά αυστηρό και έναντι των ΗΠΑ και έναντι της ε, Κίνας και για την, την επισήμανση των ε, συστατικών του παιχνιδιού και για τις χημικές ουστίες που περιέχουν. Τα, τους υδρονάνθρακες, τις, χημικές ενώσεις και με κάποιες βεβαίως, κάποια όρια ανοχής, αλλά πολύ αυστηρά. και ήταν και λογικό να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδο για να αξιολογήσουμε την ε, λειτουργία τη οδηγία. Και αναρωτιέμαι, τελικά σφάλαμε τόσο πολύ ή η επιστήμη έπεσε τόσο έξω ή εξελίχθηκε τόσο πολύ έκτοτε. Διότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σφάλματα στην οδηγία αλλά ούτε πρέπει και να τροφοδοτούμε το φόβο των πολιτών για την ασφάλεια των ε, παιδιών τους. Άκουσα με προσοχή την Επιτροπή λοιπόν και η Επιτροπή η ίδια συνειδητοποιεί ότι κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να έχουμε εδώ την ασφάλεια ότι η εποπτεία της αγοράς λειτουργεί ως σύστημα. Εφόσον λοιπόν η αγορά λειτουργεί, η νομοθεσία λειτουργεί, να ρωτήσουμε τους πολίτες γιατί ανησυχούν. Η κυρία Σαλτεμόζε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την παρουσίαση. Αν τα κατάλαβα όλα καλά βέβαια, αυτό το οποίο επιθυμείτε κύριε Επίτροπε είναι να γίνει μία μελέτη για να διαπιστωθεί κατά πόσον ε, τα παιχνίδια περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες και συγκεκριμένα τα παιχνίδια τα οποία ήταν αντικείμενο έρευνα ε, στη Γερμανία. Και πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Αν υπάρχει υποψία ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των παιδιών μα, πρέπει να δράσουμε και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Και αυτό που πάνω απ' όλα επιθυμούμε είναι πάρα πολύ γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτή την ε, μελέτη για να δούμε και να έχουμε και τη σχετική έκθεση, για να δούμε κατά πόσον ε, υπήρχαν πράγματι βάσιμοι λόγοι ανησυχία. Ό,τι αφορά τώρα τα παιχνίδια, πράγματι υπάρχουν ερευνητέ οι οποίοι μα λένε ότι δεν υπάρχουν ασφαλεί οριακέ τιμέ. Θα ήμασταν σίγουροι μόνο αν ε, καταργούνταν όλες οι ουσίες ε, οι επικίνδυνες από τα, από τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τα πλαστικά. Δεν ξέρω αν ε, ε, είναι επαρκώς αυστηροί όμως ε, οι κανονισμοί και οι οδηγίες. Πριν από 1,5 μήνα ε, μία έρευνα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής εγκρίθηκε είναι βέβαια και καθήκον των κρατών μελών να φροντίσουν ότι λειτουργούν και οι έλεγχοι στην αγορά. Από ό,τι φαίνεται, δύο μόνο είναι τα κράτη-μέλη που αποφάσισαν να υπάρξει χρηματοδότηση για τη βελτίωση των ελέγχων. Εμείς θα θέλαμε το θέμα αυτό να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης γιατί είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω να φροντίσει και η Κομισιόν να είναι στο ύψος των περιστάσεων τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε κυρία Χέντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να απευθυνθώ στον Επίτροπο Φερχόγγεν. Καταρχά είστε βεβαίω πρόσδεκτος ε, στο Κοινοβούλιο, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βρίσκεστε εδώ και καταλαβαίνουμε ότι μοιράζεστε μαζί μα την ευθύνη να μην εκθέτουμε τα παιδιά μα σε κινδύνου για την υγεία του. Θα πρέπει λοιπόν τα ζητήματα αυτά να μπορούμε να τα συζητήσουμε και μαζί σα. Επίτροπε, όταν διαπραγματευτήκατε την ε, οδηγία αυτή σε πρώτη ανάγνωση, Θυμάστε την ψηφοφορία για την οδηγία αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπήρχαν κάποιε πολιτικέ ομάδε που συμμετείχαν στι τότε συζητήσει και λέγαμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια επίπεδα ασφαλεία και για το θόρυβο και υπήρχαν μάλιστα και συγκεκριμένοι αριθμοί σε δεσιμπέλ που προτείνονταν από την αρμόδια επιτροπή και είχατε πει από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήταν πολύ ψηλή αυτή η αριθμή. Και ότι θα έχετε ένα καταπληκτικό επίπεδο το οποίο θα εξέβρεται χάρη σε επιστημονικά στοιχεία για του ε, μακρά διαρκεία και σύντομε διαρκεία θορύβου. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, τι γίνεται με τα προβλήματα ακοής που αντιμετωπίζουμε πλέον με τα παιδιά, τι γίνεται με τα πρότυπα αυτά που θα εξευρίσκονται σε αυτόν τον τομέα. Και Επίσης, για το μέγεθος των ετικετών ε, στα παιχνίδια, για την επισήμανση. Τι έγινε τελικά με την ε, επισήμανση, με το μέγεθος των αυτοκόλλητων. Πότε θα, γίνουν, ε, θα προβλεφθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ποιο θα είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για τις ετικέτες στα κίνδυνα παιχνίδια. Ευχαριστώ. Ωραία, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye και πρώτη έχει τον λόγο η κυρία Χάνσλικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό τώρα πριν τα Χριστούγεννα που ψάχνουμε δώρα για τα παιδιά. Ε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε υιοθετήσει μία καλή απόφαση για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των παιδιών αλλά πρέπει να περιμένουμε την εφαρμογή αυτών των αποτελεσμάτων που μου φέρνονται καλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Toys Show που επιτρέπει εις ε, τους ε, επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στις αλλαγές της οδηγίας. Το Νοέμβριο όμως οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφάσισαν να αποσύρουν πάρα πολλά παιδικά κρεβατάκια από τις Ηνωμένε Πολιτείε και από τα Καναδά. Ε, τα παιδιά έρχονται σε επαφή πολύ περισσότερο με τα κρεβατάκια τους από ό,τι με τα παιχνίδια. Και καλό θα ήταν η Επιτροπή να επέμβει, να εξασφαλίσει ότι είναι ασφαλή τα κρεβατάκια των παιδιών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σαφή σας λόγια και ε, ε, είναι βασικό να πούμε ότι η οδηγία ε, έχει βελτιωθεί πολύ υπέρ της ασφαλείας των παιδιών μας και ε, είναι δυνατόν να ισχύσει διεθνώς αυτή η αυστηρή νομοθεσία αλλά οι γονείς ανησυχούν, διαπιστώνουν ε, και την ε, μελέτη του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για την έρευνα και πρέπει να αναρωτηθούμε έχει δίκιο το Ινστιτούτο ή όχι διότι εν πάση περιπτώσει η κατάσταση αυτή πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ καλά διότι πρόκειται για τα παιδιά παιδιά και θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ που προθυμοποιηθήκατε να κάνετε ό,τι μπορείτε αλλά ελπίζω ότι ε, θα πάμε πιο γρήγορα. Ε, ε, είπατε μέχρι του χρόνου. Ελπίζουμε θα έχουμε τα αποτελέσματα το πρώτο εξάμεινο. Είναι βασικό να προχωρήσουμε γρήγορα για την ασφάλεια των παιδιών σας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί το Ινστιτούτο καθυστέρησε τόσο πολύ ως αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής Τι είναι ο κυριος Παπανικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιπτώσεις δεκάδων παιδιών, το 2000 μόνο ήταν 36, που χρειάστηκαν άμεση χειρουργική επέμβαση λόγω ύπαρξης βλαβερών ουσιών στα παιχνίδια. Θυμίζω επίσης ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε στην Αμερική έκθεση που αναφέρει ότι το 1 τρίτο των εγκυκλοφορία παιχνιδιών περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωση ce δεν επαρκεί ω εγγύηση ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών. η απονομή τη γίνεται έπειτα από κατάθεση σχετικού ελέγχου και του σχετικού, φακέλου από την εκάστοτε εταιρεία και όχι προληπτικού και δειγματοληπτικού ελέγχου του προϊόντο με αποτέλεσμα η ασφάλεια των παιχνιδιών να μην θεωρείται δεδομένη. για να μπορέσουν λοιπόν τα παιδιά μα δεν έχω παιδιά φιλοδοξώ όμω να αποκτήσω να δεχθούν τα δώρα του άγιου βασίλειου όπω υπόθηκε με όρου απόλυτη ασφάλεια και χωρί την ανησυχία των γονιών οφείλουμε να πιέζουμε τα κράτη μέλη για περισσότερου και πιο επισταμένου ελέγχου και βεβαίω για ενδυνάμωση τη ισχύουσα νομοθεσία. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει πάλι ο Επίτροπος Φερχόικεν. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι για την ευρεία συνένεση που ε, απεδείχθη από αυτή τη συζήτηση, αλλά έχω να πω το εξής. Έχουμε να κάνουμε ένα επιστημονικό Ινστιτούτο, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την έρευνα των κινδύνων και ε, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κινδυνολογήσει προς την κοινή γνώμη χωρίς όμως να ενημερώσουν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους για αυτή την κατάσταση των πραγμάτων. Πρέπει να σας πω ότι η, περι... περαιτέρω του Ινστιτούτου αυτό στη Γερμανία από το δημόσιο προϋπολογισμό εξετάζεται ε, αλλά δεν ε, διότι δεν ε, ε, δεν είναι χρήσιμο εάν δεν ανακοινώνει τα αποτελέσματά του. Αλλά είναι πολύ σοβαρό ακόμη και αν το διαβάζουμε στον τύπο διότι ενδέχεται να υπάρχουν νέες επιστημονικές διαπιστώσεις και ενημέρωσα την Επιστημονική Επιτροπή Δηλαδή μόλις πληροφορήθηκα ότι ενδεχομένως υπάρχουν νέες επιστημονικές διαπιστώσεις σχετικά με τις οριακές τιμές και τις επιπτώσεις αμέσως ενημερώνουμε την Επιστημονική Επιτροπή. Δεν μπορείτε όμως να απαιτείτε από μένα ή εγώ από εσά να λύσουμε τον καυγά μεταξύ των επιστημόνων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε εμείς ούτε εσείς. Μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτά τα οποία σας λέγω. Δηλαδή, να υπάρχει μία μέθοδος ε, στην μέτρηση των οριακών τιμών. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και ε, το γερμανικό αυτό Ινστιτούτο ε, εξέδωσε μία γνώμη με την οποία δεν συμφωνεί κανείς άλλος. Λοιπόν, θεωρείτε ότι εγώ θα ήμουνα υποχρεωμένος να ακολουθήσω τη γνώμη ενός μοναδικού Ινστιτούτου και όχι κανενός άλλου. Αν θέλετε πέστε μου το, αλλά εγώ δεν μπορούσα μόνος μου να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί δηλαδή, ε, δεν μπορούσα αυτοβούλος να κάνω κάτι τέτοιο. Σας είπα ότι αν υπάρξουν αντικειμενικές διαπιστώσεις θα επέμβω αμέσως. Αλλά κυρία με συγχωρείτε, κάποιος από εσά η κυρία Βάισμπεργκερ που είπε ότι θα έπρεπε να επιταχύνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα. Πρόκειται για πολύ περίπλοκα επιστημονικά θέματα, τεχνικά θέματα. Ε, κάνουμε πολλές δοκιμές σε ζώα για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε αυτές τις διαπιστώσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εν φθαλμού. Δεν είναι δυνατόν και θα πρέπει να το δεχτείτε. Αν σας λέω ότι η Επιστημονική Επιτροπή μας είπε ότι δεν μπορεί να έχει τεκμηριωμένα αποτελέσματα τα οποία θα μας δοθούν πριν από το μέσο του επομένου έτους και μόλις υπάρξουν αυτές οι νέες αποδείξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιληφθεί και θα διατυπώσει νέα νομοθετικά μέτρα. Αλλά προσπαθούμε να υπάρχει ο ελάχιστος δυνατός κίνδυνος ε, και οι ε, διαπιστώσεις μας να είναι έγκυρες. Δεν χρειάζομαι ε, άλλο για να σας τα πω αυτά. Προσπαθώ να κάνω το καθήκον μου. Κυρία Είπατε ότι θα έπρεπε να έχω απευθυνθεί νωρίτερα στον τύπο και όμως το έπραξα, θα εκπλαγείτε παρόλο που δεν πιστεύω ότι αυτά που είπα σήμερα στο Κοινοβούλιο θα επαναληφθούν ή στο γερμανικό τύπο ή στον ευρωπαϊκό κήπο διότι ε, δυστυχώς ε, δεν, δεν την επανέλαβαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση αλλά εγώ έχω κάνει τη σχετική δήλωση τύπου προκαιρού σχετικά με την πιο αυστηρή νομοθεσία του κόσμου. Μάλιστα την έχουμε κυρία και κανείς δεν μας πιάνει σε αυτό το σημείο όταν πρόκειται ιδίως για την ασφάλεια των ε, παιχνιδιών που πρέπει να είναι ε, πλήρης. Κυρία Σάλτερ Μόζερ, μπορώ να συμφωνήσω με σας. Ε, ένα κράτος δεν μπορεί να αμφισβητεί την εποπτική αρχή όσα όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής θα είναι πολύ σημαντικό και εδώ και πάλι έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα. Όσον αφορά το ερώτημα της κυρίας Χε, όσον αφορά τις προδιαγραφές, ποιες θα είναι οι προδιαγραφές για διάφορους τομείς και αναφέρατε δύο. Το ένα είναι για το επίπεδο θορύβου και πρέπει να σας πω ότι οι σχετικές ερωτήσεις έχουν υποβληθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να πετήσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει κανείς σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα ή σε λίγους μήνες να μας απαντήσουν. Χρειάζεται ο χρόνος τους. Αλλά όλα τα θέματα αυτά είναι εξελίξη και ε, ελπίζω ότι θα μας επιτρέψουν να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στα παιχνίδια τα οποία παράγονται και ε, να παρακολουθείτε και από τις εποπτικές αρχές. Ε, θα ήθελα να αναφέρω εδώ όσον αφορά τα καθίσματα των παιδιών ότι δεν πρόκειται για παιχνίδια και αναφέρονται σε διαφορετική οδηγία για την κάλυψη των προϊόντων και πρέπει να σας πω ότι το σύστημα που έχουμε στην Ευρώπη σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων βελτιώνεται συνεχώς και αν κυκλοφορούν ή βρεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που δεν είναι ασφαλή να είστε βέβαιος ότι αμέσως ενημερώνονται όλα τα κράτη-μέλη μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φερχόγγεν. Κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη συνεδρίαση θα ξεκινήσει αύριο 3η 15 Σεπτεμβρίου από τις 9 έως 1, από τις 3 έως τις 7 ε, και στις 9 έως τις 12. Παρακαλώ μπορεί